Um, Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη ερώτηση είναι η παριθμό 18 της κυρίας ε, Κράτσα. Ο αρμόδιος επίτροπος για την απάντηση είναι ο κύριος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας καταρχήν. Μόλις έφτασα από το Λουξεμβούργο, όπου το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο κανονισμού για τα hedge funds και το private equity. Και σας το λέω αυτό με το που φτάνω στο Κοινοβούλιο, γιατί ναι μεν το σχέδιο είναι σχέδιο γιατί περιμένουμε την στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το σχέδιο οφείλει πολλά στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον εισηγητή του Κοινοβουλίου, τον κύριο Γκοζές. Και πολλά από τα συμπεράσματα της ε, τελικής ψηφοφορίας ε, του Συμβουλίου και πολλά στοιχεία περί εποπτείας περιλαμβάνουν προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεργαζόμαστε στενά τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα οριστικοποιήσουμε αυτή την ε, έκθεση για τα hedge funds και το private equity. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Η κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλου μου έθεσε ερώτηση για τις συζητήσεις περί βασιλείας που έχουν σχέση με την σχετική ρύθμιση για, τη, για τα κεφάλαια της στάθμης Κιδίνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Και εδώ θα ήθελα να επενέσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του και για την θαυμάσια έκθεση του κυρίου Κάρας που πριν από δύο εβδομάδες είχαμε συζητήσει και μάλιστα θα ασχοληθείτε με την πρόταση ΣΕΡΔΕ4 που θα υποβάλουμε την άνοιξη του 2011 για να εφαρμόσουμε την Συμφωνία Βασιλεία 3 και στην Ευρώπη. Η οικονομική κρίση δεν έχει περατωθεί ακόμη, ήταν άνευ προηγουμένου και οι απώλειες, οι ζημίες των τραπεζών ήταν ε, 2-3 εκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια με βάση τους απολογισμούς του 2010. Για τις μισές από τις ευρωπαϊκές τράπεζες η κρίση αυτή βήθησε την ευρωπαϊκή οικονομία σε πολύ σοβαρή κρίση. Το ΑΕΠ το της Ευρώπης ε, ε, συρρυκνώθηκε 5%, 700 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για μία και μόνο χρονιά. Αν πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ώστε με το δανεισμό να τροφοδοτούν την οικονομία, την απασχόληση. Γι' αυτό χρειάστηκαν κάποια κατεπήγοντα μέτρα, άνευ προηγουμένα από τα κράτη-μέλη, που τότε χρηματοδοτούνταν από το φορολογούμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμ, για 4-3 και 35% του κοινωτικού προϋπολογισμού πρόβλεψε κάποια μέτρα προκειμένου να ε, βοηθήσουν βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ξεφύγουν από την κρίση και να μειώσουν τα δημόσια χρέη τους ο φορολογούμενος που πλήρωσε μία φορά θα πρέπει να συμβάλλει και δεύτερη φορά για να πληρωθούν τα σπασμένα. Όχι, κατά τη γνώμη μου, κάτι θα ήταν άδικο, γιατί η πολιτική μας ε, θα πρέπει να τάσεται υπέρ της πρόληψης. Η πρόληψη είναι φθηνότερη από την ε, διόρθωση και τη θεραπεία. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν ε, να έχουμε δεύτερη φορά τα αποτελέσματα της κρίσης. Θα πρέπει να είμαστε προνοητικοί στις πολιτικές μας θα πρέπει να εφαρμόσουμε την πρόληψη και τα μέτρα της Βασιλείας 3 ουσιαστικά εφαρμόζουν αυτή την προσπάθεια πρόληψης για την διευθέτηση των τραπεζικών κρίσεων και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να στηριχθούμε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ε, κυρίας Φερέιρα. Το G20 στον Απρίλιο του 2011 έθεσε στην, ε, στην Επιτροπή της Βασιλείας 2 να εμβαθύνει στους κανόνες και να υποβάλει νέες προτάσεις για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών και να βελτιωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Βέβαια, στις 19 και 20 Μαρτίου εγκρίθηκαν αυτές, αυτοί οι στόχοι και αναπτύχθηκαν στην Επιτροπή της Βασιλείας 2 οι προτάσεις για τη Βασιλεία 3 με τη συμμετοχή υπηρογνωμών από πολλές χώρες και την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούσε τα κράτη-μέλη. Η ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Επιτροπή Βασιλεία δείχνουν ότι οι νέοι κανόνε θα ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα μειώσουν ε, την επισφάλεια και θα καταλήξουν σε πολύ σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη για πολλούς δικαιούχους, χάρη στη μείωση της συχνότητας των τραπεζικών κρίσεων. Χάρη στην ε, μεταρρύθμιση αυτή θα ε, ενισχυθούν και οι δανειολήπτες και οι δανειοδότες, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες. Βέβαια τα ωφέλη αυτά θα φανούν σταδιακά χάρη στην σταδιακή εισαγωγή των νέων κανόνων και των μεταβατικών ρητρών που ανήγγυλαν οι, των, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών στις 12 Σεπτεμβρίου του 2010. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσει ρευστότητας που θα τύχουν υπό παρακολούθηση μέχρι το 2015 ε, ρωτήστε κύριε Αντιπρόεδρε αν με, τις νέους, με τους νέους κανόνες θα επιταχυνθούν οι συγχωνεύσεις μεταξύ των τραπεζών. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος της μεταρρύθμισης. Βέβαια, αν ε, μερικές τράπεζες δεν μπορέσουν εμπρόθεσμα να τηρήσουν τους κανόνες, ίσως θα χρειαστεί να συγχωνευτούν με τους εταίρους ή τους αντιπάλους, τους ε, ανταγωνιστές της. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την προστασία των καταθετών και των πιστωτών τους και θα συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας. Δεν θα πρέπει οι νέες διατάξεις να πλήξουν τις μικρότερες τράπεζες δυσανάλογα. Γι' αυτό και η Επιτροπή των Ελεκτών Τραπεζών θα ελέγξει τα μέτρα της Βασιλείας 3. Και η μελέτη αυτής της Επιτροπής έδειξε ότι οι μικρές τράπεζες ε, θα θυγούν λιγότερο από τους νέους κανόνες από ότι οι 50 μεγαλύτερες ε, τράπεζες και τραπεζικοί όμιλοι, χάρη στο μεγαλύτερο επίπεδο αρχικής κεφαλαιοποίησης των μικρών τραπεζών και ένα πλούσιο οικονομικό μοντέλο. Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και θα ήταν ευκταίο η G20 να μην ξεκινήσει τώρα ευρύτατη συνομιλία και διαβουλεύσεις για τα μέτρα της Βασιλείας 3, γιατί είναι ο καρπός ε, μακρύτατης και ισορροπημένης συζήτησης. Και τα αποτελέσματα της Συνόδου G20 είναι, δημιουργούν πλεονέκτημα για την Ευρώπη και ελπίζω όλοι να εφαρμόσουν έγκαιρα και σωστά τις, ε, τα μέτρα της Βασιλείας 3. Αυτά θα ήθελα να πω απαντώντας στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Επίτροπε, για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Ήσασταν πολύ πλήρης στην απάντησή σας προς την κυρία Κράτσα. Κυρία Κράτσα, θέλετε να δευτερολογήσετε. 30 δευτερόλεπτα. Μερίζομαι, κύριε Πρόεδρε, ε, την άποψή σας για την πληρότητα της απάντησης ε, του επιτρόπου κύριου Μπαρνιέ. Πράγματι αναφέρθηκε σε όλα τα ερωτήματα και δεν συμβαίνει πάντα αυτό με τις απαντήσεις της Επιτροπής. Ε, επιτρέψτε μου κύριε Επίτροπε να αναφερθώ ιδιαίτερα, ίσως να σας κάνω μάλλον μια συμπληρωματική ερώτηση για το θέμα της ρευστότητα των τραπεζών με την εφαρμογή της Βασιλείας 3. Πιστεύετε ότι δεν θα θυγεί άμεσα η ρευστότητα γιατί ήδη πλήττεται η αγορά από έλλειψη ρευστότητα των τραπεζών λόγω του ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά που η επιτροπή πιστεύει ότι δεν θα έχει επιπτώσει τη ρευστότητα αυτή τη στιγμή που τόσο την έχει ανάγκη η αγορά. σας ευχαριστώ. Um, uh, Έχω δύο επιπλέον ερωτήσει. Ο κύριος Ρούμπι και ο κύριος Έμκα. Äh, ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαρνιέ. Εμένα με ενδιαφέρουν οι επιπτώσει τη Συμφωνία Βασιλεία 3 στην Αμερικανική αγορά, όπου πολλέ μικρέ τράπεζε, εκατοντάδε, πτώχευσαν και οι μεγάλε τράπεζε. Τι έγινε με τι μεγάλε τράπεζε ε, στην Αμερική ε, πώ ακριβώ ε, εφαρμόζεται η Βασιλεία 3. Εφαρμόζεται εκεί η συμφωνία όπως και στην Ευρώπη. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα και το πρόγραμμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Βασιλεία 3 στην Αμερική. Ο κύριος Ζέμκα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση, μια και δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη ε, και η οικονομική κατάσταση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ευτυχώς ε, διαπιστώνουμε και εδώ, χάρη σε αυτή την ανησυχία, και τη φροντίδα μια βελτίωση της κατάστασης. Η ερώτησή μου είναι σύντομη. Είπατε ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια θα είναι η ουσία, η ουσία αυτών των προτάσεων που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη του 2011. Κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου κάνετε μία ερώτηση για τη ρευστότητα. Η δημοσιονομική, η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι οι τράπεζες ε, οι οποίες είχαν υπερβολική ρευστότητα δεν πήραν δάνεια. Γιατί ακριβώς ήταν πολύ συνετές, ε, κάλυπταν τις ανάγκες τους με την επαρκή ρευστότητα. Ε, όμως υπήρχε ένα έλλειμμα κατανόησης της ε, κατάστασης της υγείας των άλλων χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Νομίζω ότι νέε προτάσεις θα βοηθήσουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τη βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου για την ρευστότητα των τραπεζών, με την ενδυνάμωση των αποθεμάτων ρευστότητας. Οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπει η Επιτροπή Βασιλείας προβλέπουν ότι η νέα, το νέο επίπεδο κάλυψης ε, θα γίνει υποχρεωτικό από το 2015, κυρία Κράτσα. Αυτό θα δώσει αρκετό χρόνο στις τράπεζες, ούτω ώστε να συμμορφωθούν και να μειώσουν, ελπίζω, τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην αγορά για την μεταβατική αυτή περίοδο. Κύριε Ρούμπικα, Αναφερθήκατε στη Βασιλεία 2. Για τις Ηνωμένε Πολιτείε μιλήσατε συγκεκριμένα. Η Βασιλεία 2 δεν έχει εφαρμοστεί. Ούτε η Βασιλεία 2,5. Μάλιστα, ε, ήρθα σε συμφωνία με τον ε, Αμερικανό Υπουργό, ούτως ε, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψής μου στην, ε, στη ΣΥΠΑ, ε, έγινε η πρώτη επίσκεψη τη 9-10 Μαΐου. Ε, θα ξαναεπισκεφθώ της Αμερικής. Ε, την Βασιλεία 2,5 θα τη θέσουν σε εφαρμογή οι Αμερικάνοι το 2011. Η ερώτησή σας όμως είναι πολύ σημαντική. Γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια διεθνής δέσμευση. Οι Αμερικανοί και αυτοί δεσμεύτηκαν για να εκπονήσουν και αυτοί τους δικούς κανόνες Βασιλείας. Είναι σε μια αντίστοιχη διαδικασία. Είναι παρόντες. Επομένως είναι φυσιολογικό οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού να εφαρμοστούν από κοινού, παράλληλα. Το λέω με μεγάλη προσοχή αυτό το πράγμα. Ε, θα γίνουν παράλληλες ενέργειες με τους Αμερικανούς και στα πλαίσια της δεύτερης επίσκεψής μου θα το επαληθεύσω. Γενικά τώρα, σε ό,τι αφορά την επίπτωση στις μεγάλες ή μικρότερες τράπεζες της ε, Βασιλείας 3, θα προσέξουμε, χωρίς να κάνουμε ταχυδακτηλουργίες, και θα κάνουμε μελέτες επιπτώσεων μακροοικονομικές και μικροοικονομικές και θα χρησιμοποιήσω όλα τα περιθώρια ευελιξίας που έχουμε, ούτω ώστε να εκπονήσουμε τα κατάλληλα μέτρα να πάρουμε τις, και να παράγουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Κυρία Σέμκε, για το χρονοδιάγραμμα μου κάνετε μια ερώτηση. Αυτό που θα κάνουμε την Άνοιξη 2011 είναι να υποβάλουμε ένα σχέδιο ε, οδηγίας που θα εφαρμόσει μετά από όλες αυτές τις μελέτες επιπτώσεων, μετά από όλα αυτά τα μέτρα βαθμονόμησης ας πούμε, της ε, Βασιλείας, θα δούμε τον παραλληλισμό με άλλα μέτρα εποπτείας εσωτερικής και εξωτερικής, ε, ούτως ώστε να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα εφαρμογής της πρόληψης κινδύνου και θα υπάρξει και μια βαθμονόμηση διατλαντική. Χρειαζόμαστε κάποιους μήνες για να γίνει σωστή η δουλειά. Ε, θα ακούσουμε το Κοινοβούλιο, θα ακούσουμε τους ε, φορείς ε, του κλάδου και θα κάνουμε, θα κάνουμε προτάσεις, καλές προτάσεις ελπίζω, την άνοιξη του 2011. Θα υποβάλουμε δηλαδή νομοθετικά κείμενα. Ευχαριστούμε, πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα περνάμε στην ερώτηση παριθμών 19 του κυρίου Σαλόμ. Αφορά στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής για την επιστημική ασφάλεια και θα απαντήσει ο κ. Πίπαουλ. Φόσον μπορεί βέβαια, μόλις καθίσει στη θέση του. Και έχετε το λόγο, παρακαλώ. Το μικρόφωνο πρέπει να ανοίξετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ερώτηση αυτή θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και ε, επισητισμό. Αυτό είναι βασικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να μειωθεί κατά το ίμιση ο αριθμός εκείνων που έχουν ανάγκη. Ο πρώτος στόχος σχεδιτίας είναι μια υπόσχεση μέχρι το 2015 ε, να έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η επιστημική ασφάλεια παραμένει πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της με την Αφρική. Πολλές ε, χώρες ε, δεν ε, έχουν κατορθώσει να επιτύχουν αυτό το στόχο. Πάνω από 70% ζουν σε αγροτικές περιοχές και περίπου το 90% της γεωργικής παραγωγής ε, γίνεται σε αγροτικές, οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η επισητιστική ασφάλεια ήταν η πρώτη προτεραιότητα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Αυτή είναι και μια προτεραιότητα στους στόχους της χιλιετίας. Εμείς θέλουμε να παραμείνει προτεραιότητα στο επόμενο πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται. Επίση, επιθυμούμε να διασφαλίσουμε στοιχεία ε, που έχουν με την επιστημιστική ασφάλεια, όπω η έρευνα, το εμπόριο και η περιφερειακή ενσωμάτωση, αυτά να ε, συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα τη χιλιετία η ε, επιστημονική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζει με τη σημασία που αποδίδουν και οι ίδιοι οι Αφρικανοί ηγέτες στην επιστημιστική ασφάλεια. Ε, το πρόγραμμα ανάπτυξης της Αφρικής ε, είναι ένα κοινό πλαίσιο δράσης σε αυτόν τον τομέα και εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε αρκετούς μηχανισμούς για να λάβουμε υπόψη μας την διατροφή και την επιστημιστική ασφάλεια δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε μια νέα ε, ε, συνεργασία με την Αφρική για αυτό το θέμα. Γιατί όπως σας είπα η διάσταση αυτού του θέματος καλύπτεται ήδη ε, στη συνεργασία που έχουμε για τους στόχους της χιλιετίας και σε άλλες μορφές συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαλόμ, έχετε το λόγο για συμπληρωματική ερώτηση εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ερώτησή σας που θα είναι πολύ χρήσιμη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Μήπως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και για το είδος της συζήτησης ε, που έγινε στην ε, συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Νέας Υόρκης για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας ό,τι αφορά την επιστηστική ασφάλεια και η Επιτροπή Επιστηστικής Ασφάλειας της ΦΑΟ έτυχε της ε, δέουσας ενθάρρυνσης ώστε να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας παγκοσμίω. Ο κύριος Παπα-Νικολάου θα υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση και μετά ο κύριος Ταραμπέλα. Πριν από ένα περίπου χρόνο, τον Αύγουστο του 2009, η Επιτροπή εγκαθίδρυσε τον μηχανισμό FLEX για τις ευάλωτε χώρες δεσμεύοντα ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις πιο επισφαλείς χώρες της αφρικής για τη χρονική περίοδο. περίοδο 2009-2010. έχουμε κάποια αξιολόγηση για το πρόγραμμα αυτό ε, από την επιτροπή αν τα χρήματα αυτά πιάσαν τόπο θυμίζω ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι λαμβάνουν λιπάσματα και σπόρους για σπορά ώστε μακροπρόθεσμα να αυξήσουν τη γεωργική παραγωγή για να επιτύχουν μεσοπρόθεσμη επισητιστική ασφάλεια. σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, οι ε, πραγματικέ ερωτήσει πρέπει να είναι το μακατομέγιστο 30 δευτερόλεπτα. Πέρα από τα νούμερα που ανέφερα ο κύριο Σαλόμα, στην ε, υποσαχάρια Σαχάρα, περίπου 800 εκατομμύρια, Αφρική συγγνώμη, ζουν ε, με γεωργική παραγωγή η οποία ε, πολλαπλασιάστηκε ε, κατά 2,6. Προχώρησε πολύ περισσότερο τα τελευταία 50 χρόνια παρά τα τελευταία 10.000 χρόνια. Το... Δεν έχει νόημα στην Πουρκίνα Φάσο ας πούμε, να καλλιεργείται μόνο βαμβάκι όταν το 49% του πληθυσμού πεινάει. Δεν θα πρέπει να θέσουμε το, την επιστημιστική ασφάλεια στην, στο κέντρο της αναπτυξιακής πολιτικής. Κύριε Επίτροπε, έχετε λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, πολύ σύντομα ε, όσον αφορά την ερώτηση του κ. Σαλόμ για την συνάντηση κορυφή για του στόχου χιλιετία, νομίζω το βασικό αποτέλεσμα αυτή τη συνάντηση κορυφή είναι μια ξεκάθαρη συμφωνία ανάμεσα αναπτυγμένε και τι αναπτυσσόμενε χώρε μέχρι το 2015 να επιτύχουν του στόχου τη χιλιετία, κυρίω των υπαριθμών 1, που αναφέρει να μειωθεί η παγκόσμια φτώχεια κατά το ίμιση και να ενισχυθούν θέματα επισητιστική ασφάλεια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να λάβουμε μέτρα για να επιτύχουμε του στόχου τη χιλιετία την ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε, έχουμε δύο εργαλεία. Το πρόγραμμα Flex αφορά τις χώρες σε κρίση. Έχουμε και αυτό το πρόγραμμα ε, που έχει ως στόχο να στηρίζει τις μικρές καλλιέργειες, τους μικρούς καλλιεργητές και είχε μεγάλη επιτυχία για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Σε πάρα πολλές χώρες βελτιώθηκε η κατάσταση ως προς την επισητιστική ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο ε, μία φορά και τέλος ενώ η κρίση συνεχίζεται. Για να περάσουμε στην ερώτηση του κ. Ταραντέλα, πράγματα, η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα από τα θέματα που θα προτείνουμε στην Πράσινη Βίβλο ως ε, ένα συγκεκριμένο στόχο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όσον αφορά την, ε, τα εργαλεία. Είχαμε πολύ θετική εμπειρία, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε παραγωγική ανάπτυξη που θα βασίζεται ε, στην γεωργική δομή η οποία εξακολουθεί να επικρατεί στην Αφρική. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τον Επίτροπο και τους συναντέλφους και πάμε τώρα στην ερώτηση υπαριθμών 20 του κ. Ταραμπέλα. Ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών, έλεγχος του σεβασμού των δικαιωμάτων των επιβατών τις αεροπορικές και συνδρομικές μεταφορές. Σε αυτήν την ομάδα έχουμε 10 ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνω στους συναδέλφους που μας ακούν από τα γραφεία τους και δεν είναι παρόντες εδώ να γνωρίζουν ότι θα βρεθούμε υποποίηση να φτάσουμε σε ερωτήσει 22-23 και τις εκείνες που ακολουθούν. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ε, ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Κάλλας. Κύριε Κάλλας, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, όπως ε, επισημάνθηκε η ε, οδηγία 1371 κάθετος 2074 και ο κανονισμός 261 κάθετος 2014 για τα δικαιώματα των επιβατών ε, επισημένονται τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία όταν ε, ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Εκεί υπάρχει αναγνώριση δικαιωμάτων, ελάχιστων δικαιωμάτων πολιτών όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή με σιδηρόδρομο. Και αυτά τα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται από ειδικά γι' αυτό ορισμένους φορείς, οι οποίοι καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι γίνονται απόλυτα σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών. Το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εποπτεύει έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο σωστά στα κράτη-μέλη. Εξάλλου, οι οργανισμοί εφαρμογής δεν υποχρεούνται να αναφέρονται ε, με βάση τον κανονισμό. Απαντούν στις ερωτήσεις της ε, Κομισιόν στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τους ε, θεσμούς, κάτι που έχει κατοχυρωθεί στη συνθήκη. Σε σχέση με την κρίση ε, για ε, την ηφαιστειακή κρίση που είχαμε πρόσφατα ανταποκρίθηκε η Κομισιόν ταχύτατα ως προς την ηφαιστειακή τέφρα. Τα δικαιώματα των επιβατών πράγματι έγιναν σεβαστά με έναν αρμονικό τρόπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτύχει το στόχο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει ε, ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές και τις έχει συμφωνήσει με τις εθνικές αρχές. Είναι σε στενή επαφή και με τις εθνικές αρχές και με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Σας ευχαριστούμε. Πριν από λίγο σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τριών επιτρόπων και θα αφιερώσουμε 20 λεπτά σε ερωτήσεις προς τον καθένα. Άρα τέσσερις ερωτήσεις προς κάθε επίτροπο θα προλάβουμε να θέσουμε. Ελπίζω να φτάσουμε στην ερώτηση 23 του κυρίου Χίγκης προς τον κύριο Κάλλες. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει το λόγο για συμπληρωματική. Κύριε Πρόεδρε, Αντιλαμβάνεστε κύριε Επιτροπέ ότι η υιοθέτηση του κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών σε αεροπορικέ, αεροδρομικέ και πρόσφατα θαλάσσιε μεταφορέ ε, έγινε εύλογε προσδοκίε προ το επιβατικό κοινό ότι θα βρεθούν ε, οικονομικέ αντισταθμίσει για τι καθυστερήσει, ακυρώσει ε, και άλλα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά οι αιτιάσει του και οι προσφυγέ έχουν μείνει χωρί ε, συνέχεια. Μετά την ηφαιστειακή ε, τέφρα τη Ισλανδία. δεν αποζημιώθηκαν οι επιβάτε. Πρέπει λοιπόν να υποχρεώσουμε τι αεροπορικέ εταιρείε να εφαρμόσουν του κανονισμού και να ανάγκη να επιβληθούν και κυρώσει. Το Φεβρουάριο του 2006 στο Βέλγιο αυτές οι ρυθμιστικές αρχές δεν ε, επέβαλαν κανένα πρόστιμο στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματα των καταναλωτών. Ο κύριος Κούσα και μετά ο κύριος Παλέτσκης. Μία σύντομη ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, τι πιστεύετε για τη διαφορετική προσέγγιση στις, των διαφόρων μέσων μεταφοράς ό,τι αφορά τα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Ποιες είναι οι ιδέες ε, και ποια είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τα διάφορα είδη μεταφορών, δηλαδή εναέριες, ε, οι συνδρομικές μεταφορές δεν θα πρέπει να, έχουν, να οδηγούν σε κοινέ δέσμες ε, δικαιωμάτων και ενιαίους ελέγχους σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση με το ηφαίστειο έδειξε ότι ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά οι νέες χώρες, δεν έχουν εναλλακτική λύση και δεν υπάρχουν ε, πραγματικές συνδέσεις ε, με την Δυτική Ευρώπη. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η δική σας χώρα και η δική μου χώρα. Αυτή η κατάσταση ε, έχει επιταχύνει τις εργασίες για την Βαλτική και το σιδηρόδρομο της Βαλτικής, επίτροπε. Για την εμπειρία μας από το ηφαίστειο και την κρίση που προέκυψε με τα δικαιώματα των επιβατών. Έχουμε πλήρη μέτρα ε, και έχουμε κείμενα που μας έδειξαν ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ε, συμπεριφέρθηκαν ε, λελογισμένα, το ίδιο και οι επιβάτες. Τα περισσότερα προβλήματα λοιπόν έχουν επιληθεί. Υπάρχουν βέβαια πάντα αξιώσεις και πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν μιλάει για ακυρώσεις ε, προς τις αεροπορικές εταιρείε. Το θέμα είναι να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις αξιώσεις που δεν έχουν, στις οποίες δεν έχει δοθεί συνέχεια. Είμαστε σε επαφή με τις εθνικές αρχές και με τους εθνικούς φορείς ε, εφαρμογής ε, των κανόνων. Ε, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι άσχημη, μπορώ να σας πω. Για τη δεύτερη ερώτηση. Ναι, θέλουμε να υπάρξουν τελικά εναρμονισμένοι κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα κάνουμε μία διαβούλευση για να συζητήσουμε με το Συμβούλιο ένα προβληματικό σημείο για τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, στα Πούλμαν. Ε, και για τις εναέριες μεταφορές και για τις συνδρομικές μεταφορές θέλουμε πραγματικά μια εναρμονισμένη φιλοσοφία. Για το συνδρόμο της Βαλτικής θα κάνω ό,τι μπορώ για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να έχω τη συνεργασία τη δική σας ε, και τη συνεργασία των χωρών που τις αφορά. Ελπίζω λοιπόν η ιστορία αυτή να τελεσφορήσει. Ωραία. Ερώτηση 21 της κυρίας Χάρκιν. When you're ready, Ο κύριος Κάλλας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Μετά την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει τελικά την πρότασή της. Μια και η οδηγία καλύπτει πια και τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ε, ότι τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τους ε, κανόνες και στους αυτοαπασχολούμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη την εσωμάτωση της οδηγίας ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους ε, οδηγούς και θα αποφασίσει για ενδεχόμενα μέτρα μετά τη λήψη των απαντήσεων από τα κράτη-μέλη και την ε, επεξεργασία φυσικά αυτών των απαντήσεων. Η κυρία Χάρκιν, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Διερωτώ με, υπάρχουν προτάσεις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να ελέγξουν καλύτερα το χρόνο, το ωράριο εργασία των αυτοαπασχολούμενων, ιδιαίτερα το χρόνο που αφιερώνουν στον καθαρισμό τον, ε, ή τη συντήρηση των οχημάτων του ή τι διοικητικέ διατυπώσει, γιατί θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί αυτό. Ποιο είναι ο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο προ αυτοαπασχολούμενου, μια και το ωράριο εργασία του θα μειωθεί σημαντικά με την εφαρμογή τη οδηγία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε προτάσεις για τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Από νομική άποψη πάντως, οι διατάξεις της οδηγίας αυτής ισχύουν και θα πρέπει να τηρηθούν. Ως προς τι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα αναλύσουμε πρώτα τις απαντήσεις που θα μας στείλουν τα κράτη-μέλη και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ερώτηση 22 του κυρίου... Μάλλον, συγγνώμη, ερώτηση 23, λέει ο πρόεδρο. Όχι, λάθο. Επανέρχεται στην ερώτηση 22 του κυρίου Κομουτσάκου και ερώτηση 23 του κυρίου Χίγκινς για ειδικά μέτρα για τα σχολικά λεωφορεία και τους οδηγού του και την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος Κάλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι ε, είναι μεγάλος ο αριθμός των, τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Το 2009 35.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σαν να χάθηκε δηλαδή μια μικρή κομμόπολη, ο πληθυσμός μιας κομμόπολης. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει το τρίτο πρόγραμμα δράσης 2001-2001 που δυστυχώς είχε αποτύχει Είχαμε βέβαια μια κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μωρών, μερών και κατά την περίοδο αυτή 78.000 ζωές σώθηκαν στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 2 εκατομμύρια θύματα. Σώσαμε πολλές οικογένειες και γλιτώσαμε πολλές οικογένειες από φοβερή οδύνη και είναι ανεκτήμητες αυτές οι προσφορές. Σε ό,τι αφορά την ε, το πρόγραμμα δράσης για την ειδικη ασφαλεια ασφάλεια 2011-2020 θα συνεχίσουμε την υλοποίηση των στόχων του περιορισμού των ε, θανατηφόρων τροχαίων και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα του 2010. Φυσικά για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ε, θα απαιτήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και από τα κράτη-μέλη και πιο ισχυρή ανάμειξή τους, ε, ιδιαίτερα από τα κράτη που έχουν τις χειρότερες επιδόσεις στα τροχαία. Ελπίζω να δημιουργηθούν αποτελεσματικές εθνικές στρατηγικές, αξιοποιώντα βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Επίσης, θα πρέπει να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, ιδιαίτερα με τις μοτοσικλέτες ή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ε, επαρχιακών οδών. Θα πρέπει να αναπτύξουμε και ευφύστηματα μεταφορών, γιατί ο δικό του ρόλο θα είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση των στόχων μα. Σε ό,τι αφορά το ειδικό θέμα τη πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων με συμμετοχή παιδιών, ιδιαίτερα στα σχολικά λεωφορεία, σημειώνουμε την εντυπωσιακή πρόοδο που σημειώθηκε την προηγούμενη δεκαετία με τη μείωση κατά 70% του αριθμού μοιραίων ατυχημάτων με παιδιά ε, νεότερα το 15 χρόνο. Φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασία των παιδιών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού, των χρηστών ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Κουμουτσάκο, πρώτα και μετά από τον κύριο Χίγκινς. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Επίτροπε για την απάντησή σας. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνω στην ερώτησή μου γιατί κύριε Επίτροπε κάθε μέρα εκατομμύρια μαθητέ πηγαίνουν και φεύγουν από τα σχολεία του με οχήματα που χρησιμοποιούνται ως ε, σχολικά λεωφορεία. μιλάμε κυριολεκτικά για το άνθος της ευρωπαϊκής νεολαίας και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πιο αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για αυτά τα οχήματα πιο αυστηρούς και συχνούς ελέγχους για το αν εφαρμόζονται αυτά τα standards και οπωσδήποτε πιο αυστηρό έλεγχο για τις επαγγελματικές ικανότητες των οδηγών αυτών των λεωφορείων. κύριε επίτροπε νομίζω ότι θα πρέπει η επιτροπή να εξετάσει μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει πολύ θετικά αποδεκτή και από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη διότι μιλάμε όπως σας είπα για μια πολύ ευπαθή ομάδα που αγγίζει και το μυαλό και τις καρδιές όλων των ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ με τον Επίτροπο. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις επιδόσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί μόνο το 2009 έχασαν τη ζωή τους 35.000 άνθρωποι σε τροχαία ατυχήματα. Και είχαμε 15.000 ε, θύματα περισσότερα από τον αρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τελευταία περίοδο. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο, υπάρχει κάποια πρόταση για ενίσχυση αυτού του σχεδίου δράση, γιατί δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Θα ακούσουμε δύο ακόμη συμπληρωματικέ ερωτήσει από την κυρία Τσικάου και την κυρία Χάρκιν. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεδομένου ότι είχαμε 35.000 θύματα σε μοιραία τροχαία ατυχήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι σαν να χάνουμε μία μικρή πόλη κάθε χρόνο από το χάρτη εξαιτία των τροχαίων ατυχημάτων. Το 50% των θυμάτων είναι πεζοί, ποδηλάτες ή μοτοσυκλετιστές. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε μία ε, σωστή διαπαιδαγώγηση ήδη από το σχολείο και να ενημερώσουμε τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού με κατάρτιση ήδη από τα σχολικά χρόνια. Κυρία Χάρκιν, σε ό,τι αφορά τα σχολικά λεωφορεία, η Επιτροπή έχει σκεφτεί την πρόταση όλα τα παιδιά κατά να δένονται με ζώνη ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία και μόνο ένα παιδί να κάθεται σε κάθε θέση. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά λεωφορεία, ισχύουν πολύ αυστηρέ διατάξει για τι τεχνικέ προδιαγραφέ που θα πρέπει να πληρούνται από τα σχολικά λεωφορεία. Δεν έχω ακούσει ιδιαίτερε ανησυχίε για σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα με τα σχολικά λεωφορεία ή τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται ω σχολικά. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και Θέλουμε να εφαρμοστούν αυστηρά οι κανόνες. Θα πρέπει να κάθονται σωστά όλα τα παιδιά, να μην στριμώχνονται στις θέσεις και φυσικά να δένονται με ζώνες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν επισημανθεί ιδιαίτερε ανησυχίες εις βάρος των σχολικών λεωφορείων στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια. Είναι όντως ε, μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, 30.000 και, και κάθε θάνατος είναι μια τραγωδία. Δεν συμφωνώ όμως ότι το σχέδιο δράσης για την οδική ασφάλεια ήταν αποτυχημένο. Γιατί οδήγησε σε μείωση κατά 40% των μοιραίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Και τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια είχαμε ε, υποτετραπλασιασμό στην δική μου πατρίδα των μοιραίων ατυχημάτων. Πριν τις θερινές διακοπές υιοθετήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια και στόχος μας είναι να μειώσουμε τα τροχέα στο ίμιση. Επίσης θα υποβάλουμε μέτρα προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η κατάρτιση η ενημέρωση και η σωστή διαπαιδαγώγηση των πιο ευπαθών στρωμάτων του πληθυσμού. Και φυσικά οι πιο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσυκλετιστές. Αυτά τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί οι μοτοσυκλετιστέ ήταν η μόνη κατηγορία στου οποίου τα μοιραία ατυχήματα αυξήθηκαν, ενώ όλε οι υπόλοιπε κατηγορίε μειώθηκαν. Ευχαριστώ. Πάμε στην ερώτηση 24 του κυρίου Παλέκης για την υπερβολική ναυσιπλοεία στη Βαλτική θάλασσα. Θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. It's question 24. Παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτηση 24. Στα δικά μου χαρτιά έχω άλλα νούμερα. Αλλά το ερώτημα του κυρίου Παλέκης μπορώ να το απαντήσω. Λόγω της ε, ταχείας οικονομικής ανάπτυξης αυξάνονται οι μεταφορές ε, στη Βαλτική θάλασσα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα ε, έχει ένα πολύ προηγμένο πλαίσιο για την, την ασφαλή ναυσιπλοεία. Από τα πιο ασφαλή στον κόσμο σήμερα τρίτο πακέτο για την αυσιπλοεία που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2009 είναι μια σημαντική βελτίωση ε, για την παρακολούθηση, για την καταγραφή, καλύπτει όλη τη θάλασσα γύρω από την Ευρώπη και εισάγει αυστηρές επιθεωρήσεις στα πλοία που επισκέπτονται ε, τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη Βαλτική, όπως παραδείγματος χάρη ασφαλής ναυσιπλοεία και ασφαλή πρότυπα για τους πάγους. Επίσης υπάρχει πρόνοια για την ε, καλή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Υπάρχει και τεχνική υποστήριξη από την ε, Υπηρεσία Ναυσιπλοείας. Αν υπάρξει ατύχημα, η ΕΜΣΑ έχει ε, την ευθύνη ε, για να κρατήσει ε, ακινητοποιημένο το πλοίο. Αυτό επιπροσθέτω συγγνώμη, από τα μέτρα που έχουμε πάρει για τη ρήπανση, κυρίως στα βαλτικά κράτη. Ε, θέλουμε τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν ενιαία στη Βαλτική θάλασσα, γι' αυτό έχουμε διάλογο με την Ρωσική Ομοσπονδία η ε, Επιτροπή θα ε, ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για, την θαλάσ... για τις μεταφορές στη Βαλτική. Πρόσφατα υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ασφάλεια και της Βαλτικής. Ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση για τη μείωση των θαλασσιών μεταφορών στην ε, Βαλτική. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε περιορισμό στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να εξεταστεί πριν εισαχθεί προσεκτικά. Και θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με το δίκαιο του ΟΗΕ για το δίκαιο στη θάλασσα και τις υπόλοιπες διεθνείς συμβάσεις, καθώς ε, και τα όσα προβλέπει η Διεθνής ε, Οργάνωση Ναυσιπλοείας. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των ατυχημάτων και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σχετικά φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο μέσω μεταφοράς. Πέρα από τους περιορισμούς ε, στις μεταφορές ε, στη Βαλτική, αν προβούμε σε ένα τέτοιο περιορισμό, μπορούμε να προωθήσουμε άλλες μεταφορές που είναι λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικές και μπορεί να, αυξηθεί έτσι, να αυξηθούν έτσι και οι εκπομπές. Κάτι που δεν το επιθυμούμε. Ο κύριος Παλέκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τη λεπτομερή και πιστική σας απάντηση. Χάρηκα που άκουσα να μιλάτε για την συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι για τα πρότυπα των πλοίων για να υπάρξει περιβαλλοντική βελτίωση, πρέπει να δούμε ποιες χώρες ε, είναι καλύτερες στον τομέα αυτό, ποιες χώρες δίνουν το παράδειγμα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ, Επίτροπος. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Δεν έχω στοιχεία να σας πω ότι η τάδε χώρα είναι καλύτερη από τη Δίνα. Γενικώ πώς οι χώρες της Βαλτικής όλες είναι πολύ ευαισθητοποιημένε στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα θαλασσιών μεταφορών. Ξέρετε ότι οι σκανδιναβικές χώρες ξεκίνησαν κάποια μέτρα για να μειώσουν το θείο στα καύσιμα των πλοίων και στις εκπομπές επομένως των ε, πλοίων. Δεν έχω στοιχεία λοιπόν για να μπορέσω να εντοπίσω ποια χώρα είναι καλύτερη από τις άλλες. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ε, είσαστε μοντέλο ε, στις απαντήσεις σας. Ε, οι απαντήσεις σας είναι σύντομες, μας βοηθάνε και είναι και πάρα πολύ ακριβείς. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις του κυρίου Τσόλος. Κοινέ απαντήσεις στις ερωτήσεις 31, 32, 33, 34 και 35. Περιμένω τον Επίτροπο να λάβει θέση. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Θα απαντήσω σε αυτές τις πέντε ερωτήσεις ομαδικά που αφορούν το ίδιο θέμα. Το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλά την ε, γεωργική παραγωγή και την μέση ενίσχυση με βάση μια ιστορική περίοδο. Λόγω του γεγονότος ότι η ιστορική αναφορά που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των άμεσων πληρωμών, αυτή η ενίσχυση διαφοροποιείται ανά κράτος μέλος ε, και ανά περιοχή και ανά κατηγορία γεωργού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 12 νέα κράτη-μέλη είναι σε φάση προοδευτική εφαρμογή αυτών των άμεσων πληρωμών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 10 οι άμεσε πληρωμές θα φτάσουν στα, στο επίπεδο του 100% το 2013. Και για τις δύο τελευταίες χώρες, δηλαδή τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα, τους, θα εφαρμοστούν προοδευτικά αυτές οι άμεσες ε, ε, πληρωμές το 2016. Θα ξεκινήσουμε με ένα επίπεδο 25%. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δηλαδή το 2007. Έτσι όλα τα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη και τα 12 έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις άμεσες πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιχορηγήσεις εθνικές μέσα στα όρια που καθορίζει ο κανονισμός και οι συνθήκες προσχώρησης. Το Συμβούλιο ε, κατά κατά τον υγειονομικό έλεγχο της ε, γεωργικής πολιτικής που ξεκίνησε το 2008 ζήτησε από την Κομισιόν να εξετάσει τη δυνατότητα εξέλιξης του συστήματος ε, άμεσων πληρωμών ε, ειδικά σε ό,τι αφορά το επίπεδο διαφοροποίησης των πληρωμών κράτος μέλος. Για την περίοδο μετά το 2013 η Κομισιόν θα μελετήσει και θα αξιολογήσει τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ε, άμεσων πληρωμών. Η ε, απαραίτητη προσαρμογή του συστήματος των ε, πληρωμών αυτών και η κατανομή τους θα γίνει έτσι ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία και ισοτιμία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ διαφορών κατηγοριών ε, γεωργών. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα που συζητείται σήμερα στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχουν παρόλα αυτά ερωτήματα σε ό,τι αφορά του τρόπου και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε ε, προ μια πιο δίκαιη κατανομή. Ένα σημαντικό ερώτημα για την μελλοντική κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών είναι το να καθορίσουμε πώς θα περάσουμε από την σημερινή κατάσταση σε μια μελλοντική πιο δίκαιη κατανομή αποφεύγοντας ε, διαταραχές, προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν ε, αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιοχές ή για ορισμένα συστήματα παραγωγής. Η ΚΑΠΑ μετά το 2013 θα πρέπει να απαντήσει σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις, ιδίως το θέμα της επιδίνωσης του, των ευρωπαϊκών εδαφών, που σήμερα είναι ένα μίσον πρόβλημα και που επιδεινώνεται περαιτέρω από την κλιματική αλλαγή. Η βιοπικιλότητα επίσης είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τη διαχείριση τη βιώσιμη των φυσικών πόρων ε, στο εσωτερικό της στρατηγικής ε, για την Ευρώπη του 2020. Ε, μέχρι το 2010 είχαμε πει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας. Αυτό δεν το πετύχαμε. Παρ' όλα αυτά έχουν σημειωθεί θετικά βήματα και η κοινή γεωργική πολιτική νομίζω ότι συνεισέφερε σε αυτήν την προσπάθεια πολύ. Σήμερα η κοινή γεωργική πολιτική υποστηρίζει την ε, βιώσιμη διαχείριση των εδαφών με άμεσες πληρωμές ε, υπό τον όρο ότι υπάρχει σεβασμός των ε, περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, κυρίως καλές γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των εδαφών, τη διαβροσή τους, την περιεκτικότητα σε οργανικά στοιχεία. Πληρώνοντας λοιπόν αυτά τα μέτρα τα γεωργοπεριβαλλοντικά, πέρα από που ξεπερνούν τις ε, καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές. Επίσης, για να υπάρχει καλή διαχείριση των ε, ευρωπαϊκών εδαφών και για να εξασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο ε, οργανικών στοιχείων, το 2006 παρουσιάσαμε μία οδηγία πλαίσιο για, την, για τα εδάφη. Ο στόχος ήταν να εντοπίσουμε τους λόγους της διάβρωσης και να την παρεμποδίσουμε. Σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα, η ΚΑΠ σήμερα αναφέρεται στο σεβασμό των περιβαλλοντικών διατάξεων και στην οδηγία για τα πτηνά, την οδηγία, καθώς και την οδηγία για τα οικοσυστήματα. Ε, προβλέπονται επίσης ε, κυρώσεις που μειώνουν τις άμεσες πληρωμές αν δεν υπάρχει σεβασμός, καθώς και μέτρα για τις ε, περιοχές Natura 2000, καθώς και για περιβαλλοντικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ μετά το 2013, η Κομισιόν γνωρίζει το εύρος των προκλήσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και μελετάμε αυτή τη στιγμή τις διάφορες δυνατότητες, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στοιχείων σε όλα τα κείμενα, σε όλα τα εργαλεία ε, τη ε, κοινή γεωργική πολιτική του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Η ανάλυση για την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2013 είναι εν εξελίξη και μια ανακοίνωση για τι κατευθυντήριε γραμμέ τη ΚΑΠ προβλέπεται το Νοέμβριο του 2000... προβλέπεται μάλλον για τον Νοέμβριο του 2010. Θα την παρουσιάσω αυτή την ανακοίνωση στην Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου στις 17 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ κύριος Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζετε τις ουσιώδεις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των επιμέρους περιφερειών και των κρατών μελών της Ένωσης στον γεωργικό τομέα. Αναφέρομαι μεταξύ άλλων στην έκταση, την ε, διάρθρωση και την τυπολογία των εκμεταλλεύσεων, στη συμβολή της γεωργίας στην απασχόληση και την οικονομία, στις μειονεκτικές περιοχές καθώς και στις περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές. για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να καθοριστεί ενιαία ενώ σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης στραματική ενίσχυση ενιαία αυτό που λέμε flat rating. Επιβεβαιώνεται, κύριε επίτροπε ότι θα αναδειχθούν αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για την απάντηση που δώσατε σχετικά με τη διάβριση του εδάφους αλλά θα ήθελα να κάνω και μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, στις μεσογειακές περιοχές ένα βασικό αίτιο είναι ότι οι υπάρχουν απογύμνωση και αυτό οδηγεί σε πυρκαγιές, ε, κάτι που χαρακτηρίζει τη Μεσόγειο. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ε, υπολογισμού έτσι ώστε να υπάρχουν συμπληρωματικά ε, πριμ για τις αγροτικές εκείνες εκμεταλλεύσεις οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν πρακτικές οι οποίες σέβονται το περιβάλλον που όμως πρώτα απ' όλα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τις πυρκαγιές και ε, στις γεωργικές περιφέρειες. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, απάντησή σας ε, στην ερώτηση. Όπως είπατε, η ε, Βουλγαρία και οι Ρουμανοί που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα στο 40% των γεωργικών επιδοτήσεων που ε, χορηγούνται σε χώρες όπως στη Γερμανία και τη Γαλλία. Είπατε ότι ε, οι ενισχύσει αυτές θα εξισορροπηθούν το 2016. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο και με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται η γεωργία. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κυρίως ε, όσον αφορά αυτές τις δύο χώρες. Κύριε Επίτροπε, αν είστε έτοιμος μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. για την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστάμκου. Όντως υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ περιφερειών και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών γεωργών. Γι' αυτό είπα κατά επανάληψη ότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών, ίδιες δηλαδή πληρωμές αναστρέμα για όλες τις κατηγορίες. Δεν είναι αυτή η λύση. Με βάση το σύστημα των ιστορικών αναφορών ε, υπολογίσαμε επιχορηγήσεις, πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό το σύστημα, θέλουμε να το αντικαταστήσουμε με αντικειμενικά κριτήρια. Ε, θα πρέπει επίσης να προσέξουμε το ώστε η επανισορρόπηση να γίνει με μεταβατικό, βαθμιαίο τρόπο, ώστε όσοι τιμωρηθούν από αυτό το σύστημα τροποντινά, να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Θα πρέπει να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια που θα συνδυαστούν ούτως ώστε να υπάρξει μια μετάβαση έτσι ανεκτή και βιώσιμη για όλους. Κύριε Λαβία, όλα αυτά τα θέματα που συζητάτε μπορούν να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του δευτέρου ε, πυλώνα ε, στα πλαίσια των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. Ε, θέλουμε να τα διατηρήσουμε αυτά τα μέτρα και να λάβουμε υπόψη μας την ιδιαιτερότητα κάποιων περιφερειών. Αυτά που, αυτές που αναφέρατε είναι περιοχές όπου υπάρχει διάβρωση, ε, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ξεκινούν οι πυρκαγιές. Τα κράτη-μέλη, μέσω του κανονισμού που θα προτείνουμε για την περίοδο μετά το 2013, μπορούν να λάβουν υπόψη αυτά τα ειδικά προβλήματα στα πλαίσια των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και να υπάρξει ένα σύστημα συγκεκριμένη ειδική ενίσχυση για αυτέ τι περιφέρειες. Ε, νομίζουμε ότι ακριβώ για αυτό το λόγο είναι χρήσιμη η ευελιξία. Ε, για να υπάρξει καλή διαχείριση των φυσικών πόρων, τόσο στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ειδικά μέσα και εργαλεία στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε ε, να λυθεί στα πλαίσια της ευελιξίας που χορηγούμε στα κράτη-μέλη. Για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία τώρα. Κατά τη διάρκεια των ε, προενταξιακών διαπραγματεύσεων για αυτά τα κράτη-μέλη ε, προβλέψαμε ένα σύστημα phasing in, σταδιακής δηλαδή αύξησης των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό προβλεπόταν από τη συνθήκη. Το 2008, κατά τη διάρκεια του υγειονομικού ελέγχου της ΚΑΠ, είχαμε πει ότι κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης για την περίοδο μετά το 2013, τότε θα λάβουμε υπόψη και αυτό το θέμα της επανισορρόπησης του επίπεδου των πληρωμών. Αυτό το θέμα λοιπόν δεν το ξεχνάμε. Θα πρέπει να βρούμε μια ικανοποιητική λύση και δημοσιονομικά, ούτω ώστε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, αν γίνεται. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση που έχω είναι του κυρίου είναι Κάντενμπερκ, η 36. Κύριε λοιπόν Κάντεμπερκ, η παριθμόν 36. Έχετε το λόγο. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι η εφαρμογή της ε, πολλαπλής συμμόρφωσης από τα κράτη-μέλη μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό τονίστηκε από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου το 2008. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η ανάλυση που έκανε το Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεση βασίστηκε σε μία περίοδο διετίας, αμέσως μετά την εισαγωγή των καλών γεωργικών ε, προϋποθέσεων και καλών περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και μέτρων. Η εφαρμογή λοιπόν την πρώτη χρονιά το 2005 της πολλαπλής συμμόρφωσης επρόθεσε διάφορες πρωτοβουλίες ε, η Κομισιόν με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να σεβαστούν τις ε, νομικές υποχρεώσεις. Η βοήθεια της Κομισιόν γίνεται μέσω πολλών ανταλλαγών επιστολών και συζητήσεων σε διάφορα φόρουμ. Ε, εκεί ακριβώς συζητάμε τα πιο εξειδικευμένα θέματα. Ε, τα αριθμιστικά τώρα ε, ζητήματα ρυθμίζονται στην Διαχειριστική Επιτροπή που είναι αρμόδια για αυτό το θέμα και οι πιο τεχνικές συζητήσεις γίνονται σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδική που ασχολείται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Οι συζητήσεις για τις τεχνικές ελέγχου γίνονται σε ένα συγκεκριμένο εργαστήρι που έχουμε προβλέψει. Επίσης, η Κομισιόν δημοσιεύει τακτικά από το 2004 έγγραφα ανατολισμού για τα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσει να προσαρμόσουν λοιπόν τα εθνικά του συστήματα. Η παρακολούθηση από την Επιτροπή των νομικών ε, υποχρεώσεων των κρατών μελών γίνεται με βάση τις πληροφορίες που διαβάζονται μέσω ελέγχων που γίνονται στα κράτη-μέλη, επιτόπου δηλαδή. Όταν ε, εντοπίζουμε σε αυτούς τους ελέγχους αδυναμίες, προβαίνουμε σε οικονομικές διορθώσεις για τις δαπάνες των κρατών μελών. Και αν εντοπίσουμε ένα κίνδυνο για το Γεωργικό Ταμείο, ε, όπω συνέβη στο παρελθόν, ε, ξεκινάνε διάφορε διαδικασίε. Ορισμένε τρέχουν ακόμα και σήμερα. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι το σύνολο αυτών των πρωτοβουλειών επέτρεψε μια σημαντική βελτίωση τη λειτουργία του συστήματο πολλαπλή συμμόρφωση, ιδίω από την εποχή που διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο ποια είναι η κατάσταση το 2007. Οι προσπάθειες βεβαίως θα συνεχιστούν γιατί η Κομισιόν θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα. Είναι σημαντικό ε, στοιχείο εκ των όνου κάνευ της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, κύριο Επίτροπο για την ε, πραγματικά εκτενή απάντησή του και θα ήθελα να έχω μία άλλη ερώτηση από την πολλαπλή δια... Ε, πάμε στη βιοπικιλότητα. Η σωστή γεωργία μπορεί να συμβάλλει στο να αναχαιτιστεί η εξαφάνιση ειδών και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο το καθήκον του αρμόδιου Επιτρόπου για το περιβάλλον το να ευαισθητοποιήσει για αυτό το θέμα. Και συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς κύριε Επίτροπο, τι θα κάνετε εσείς έτσι ώστε η πολιτική ε, ταγή να ενημερώσουν τους πολίτες, ε, να τους ε, ευαισθητοποιήσουν για την αξία της βιοπικιλότητας και για το με αυτήν συνδεόμενο σύστημα παροχής υπηρεσιών και θα ε, δεχθούμε και τη συμπληρωματική ερώτηση της κυρίας Μακίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις. Εάν υπάρχουν ε, προβλήματα με το τρέχον σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε και περισσότερα προβλήματα που θα προκύψουν ενδεχομένω στον πυλώνα 1, αν εμβαθύνουμε στην πολυπαντική πολιτική. Αυτό αναφέρεται στο έγγραφο ε, που έχει κατατηθεί σε σχέση με την κοινή πολιτική και θα ήθελα τη γνώμη σας επ' αυτού. Ο Επίτροπος. It's okay. Donc, euh, moi, ce que je constate actuellement, c'est que je... Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι οι φορολογούμενοι, οι καταναλωτές και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι οι πιο ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα και ε, απαιτούν, ε, έχουν πολλές απαιτήσει, ψηλές απαιτήσει από τους γεωργούς. Θα πρέπει όμως να δώσουμε την ευκαιρία και τα μέσα και στους γεωργούς να κοινοποιήσουν τις προσπάθειες που κάνουν ακόμη και όταν θέτουν σε εμπορία την παραγωγή τους. Και στο σύστημα ποιότητας για τα αγροτοτροφημικά προϊόντα που θα αναθεωρήσουμε, που θα μεταρρυθμίσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε την ευκαιρία και στους γεωργούς να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους καταναλωτές για τα προϊόντα τους, να τους ενημερώσουν για τις προσπάθειες που κάνουν, για όλα τα στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη για τη φροντίδα τους περί βιοπικιλότητας κτλ. Και κυρίως την ανάγκη λήψη υπόψη των διαφόρων συστημάτων γεωργικής παραγωγής. Γιατί έχουμε τέτοια ποικιλομορφία των διαφόρων συστημάτων γεωργικής παραγωγής που μας ε, κάνει να θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την, ε, αυτό τον πλούτο των διαφόρων συστημάτων γεωργικής παραγωγής και να ενθαρρύνουμε άμεσες επαφές μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, χρηστών. Θέλουμε οι γεωργοί, χάρη στο προϊόν που θέτουν σε εμπορία, να έχουν καλύτερη επικοινωνία με τους καταναλωτές και να ενημερώνουν τους καταναλωτές για όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν και όλες τις διατάξεις που πρέπει να σέβονται. Επίσης, χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο μεταξύ της γεωργικής παραγωγής και του αγροτοτουρισμού. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος για να δώσουμε την ευκαιρία στο γεωργό να ενημερώσει τον καταναλωτή για όλη την προσπάθεια που κάνει, τη φροντίδα του για το περιβάλλον, τη φροντίδα του για το τοπίο, για την ύπεθρο και πώς εντάσσεται αυτή η φροντίδα στην γεωργική παραγωγή. Όλοι αυτοί είναι στόχοι της ε, γεωργικής πολιτικής, θα ενισχυθούν στο μέλλον και θα χρησιμοποιηθούν από τους γεωργούς για να ε, ενημερώνουν καλύτερα και να βελτιωθεί η επικοινωνία τους με τους καταναλωτές για τις προσπάθειες που ήδη καταβάλουν. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτηση, κατά τη γνώμη μου, οι κανόνες και οι διατάξεις για το περιβάλλον ή για τις ε, εργασίες, τις αγροτικές εργασίες που λαμβάνουν υπόψη την χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων δεν είναι άσχετες ε, με το κοινωνικό ζήτημα και το οικονομικό ζήτημα. Στις προτάσεις που θα υποβάλουμε στις 17 Νοεμβρίου και θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια, η πρόταση δεν είναι να αποσπάσουμε την προσοχή, να τη μεταθέσουμε από το κοινωνικό-οικονομικό πεδίο στο περιβαλλοντικό. Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε καλύτερα και να εντάξουμε την περιβαλλοντική πτυχή στη μέρημνα του γεωργού, ώστε στο μέλλον πραγματικά να μιλούμε για ανταγωνιστική γεωργία. Και για να είναι ανταγωνιστικό στο μέλλον ο Γεωργός θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και από οικονομική άποψη αλλά και από περιβαλλοντική άποψη, δηλαδή για το ανάλογα με το πώς διαχειρίζεται το έδαφος, το είδωρ, τους φυσικούς πόρους, αλλά και υπό το πρίσμα της διατήρησης των θέσεων εργασίας στην Ήπεθρο. Η ενίσχυση του, της περιβαλλοντικής πτυχής της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων στην ΚΑΠ δεν σημαίνει ότι μειώνουμε την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανταγωνιστικότητα του Γεωργού ή ότι αμελούμε τις κοινωνικές πτυχές. Και μάλιστα στις προτάσεις που θα υποβάλουμε στο μέλλον θα σας δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα για την σωστή συμπερίληψη και της περιβαλλοντικής πτυχής. Περνάμε στην τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Τσόλο, στην υπαριθμό 37. Ο κύριος Χουντής θα έχει θέσει την ερώτηση για το Ταμείο Εγγύσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τους γεωργούς και Το πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης ε, για την περίοδο 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το ΦΕΟΚΑ και το Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει εγγυητικά κονδύλια για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καμία αίτηση μεταρρύθμιση του προγράμματος δεν έχει περιληφθεί προκειμένου να συμπεριληφθεί και ένα τέτοιο εγγυητικό ταμείο. Δεν έχει υποβληθεί στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι ελληνικέ αρχέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι στα πλαίσια της επικουρικότητας ε, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια να προτείνουν το περιεχόμενο των μέτρων ε, αγροτικής ανάπτυξης με βάση τον κανονισμό αγροτικής ανάπτυξης. Με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού 1698 του 2005 που αφορούν ε, την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΦΕΝΤΕΡ, τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη μπορούν να θεωρηθούν κατέτηση των κρατών μελών και μετά από έγκριση τη Εθνική Επιτροπής παρακολούθηση, μετά από εξέταση και έγκριση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τον αλληλευτικό κλάδο στην Ελλάδα, οι εθνικέ αρχέ ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεσή του να θεσπίσουν ένα νέο χρηματοοικονομικό μέσο προκειμένου να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις του αλληλευτικού τομέα. Με βάση τις ελληνικές αρχές, το χρηματοδοτικό αυτό μέσο θα ενταχθεί σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει και είναι το TEMP. Ε, Ταμείο Εγκαιδοσία Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει αυτό το μέσο μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, επιχειρησιακών για την περίοδο 2007-2013. Η θέσπιση τέτοιων μέσων προβλέπεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Αλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ τέτοιων, της θέσπισης τέτοιων μηχανισμών προκειμένου να, να εφαρμοστούν τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος αρκεί να τηρούνται οι νομικές διατάξεις και ιδίω τα άρθρα 34-37 του κανονισμού 498 του 2007. Τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας θα ανέλθουν σε 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα κριτήρια επιλογής ε, για τους δικαιούχους θα αποφασιστούν από την ε, Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι ελληνικές αρχές αυτή τη στιγμή οριστικοποιούν το σχέδιο δράσης τους που θα συμπεριλάβει και τους όρους λειτουργίας του χρηματοοικονομικού μέσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το μέσο αυτό που τη χάνει τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ελευτικό Ταμείο να τεθεί σε εφαρμογή πριν τα τέλη του 2010. Ευχαριστώ. Κύριε Χουντή, τη συμπληρωματική σα ερώτηση παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, η απάντησή σα ήταν σχεδόν πλήρη και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώ συμπληρωματικά θα σα έλεγα αν αυτή την πρόταση η ελληνική κυβέρνηση την έχει κάνει πολύ συγκεκριμένα δώσατε κάποιες ε, πλευρές της ερώτησης και αν αυτό που είπατε εξαρτάται, δηλαδή αν αυτά θα λειτουργήσουν από το 2010, εξαρτάται από κατά πόσο εγκαίρως η αίτηση θα έρθει από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει η συγχρηματοδότηση στα σημεία που αναφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να διευκρινίσω αυτό το θέμα, το ερώτημα είναι διτό. Το ένα αφορά το γεωργικό κλάδο, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου και δεύτερο σκέλος αφορούσε τον αλληλευτικό κλάδο. Αυτό που είπα στην απάντησή μου ήταν ότι οι ελληνικές αρχές δεν υπέβαλαν αίτημα για ένα αντίστοιχο μέσο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον γεωργικό κλάδο. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλαν μόνο για τον αλληλευτικό κλάδο είπα ότι για τον αλληλευτικό τομέα μετά από αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης το χρηματοδοτικό αυτό μέσο θα είναι έτοιμο για τα τέλη του 2010, ενώ για το γεωργικό κλάδο, επειδή δεν έχει υποβληθεί ακόμη επίσημα αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, δεν μπορώ να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες. Είπα ότι εναπόκειται σε διακριτική ευχαίρεια των κυβερνήσεων να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις μετά από πρόταση ίσως να τροποποιήσουν το πρόγραμμα Αγροτική ανάπτυξη ε, μετά από πρόταση τη αρμόδια ε, επιτροπή παρακολούθηση. Αλλά για τον γεωργικό κλάδο οι ελληνικέ αρχέ δεν έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Πάμε τώρα σε ερωτήσει προ την κυρία Δαμανάκη και ξεκινάμε με την ερώτηση παριθμών 40. Τώρα δεν ξέρω πόσε ερωτήσει θα προλάβουμε ε, σήμερα το βράδυ. Πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις 8.30 έτσι ε, ώστε οι διερμηνείς να μπορούν να προλάβουν να φάνε πριν επανέλθουν στις 9 η ώρα. Ε, κύριε Δαμανάκη, αν είστε έτοιμοι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, President. European Union Aquaculture στο πρόεδρε, η υδατοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι η αιχμή του δόρατος ε, της αηφόρου ανάπτυξης. Η Κομισιόν πρέπει να ομολογήσει ότι ο τομέας της ε, υδατοκαλλιέργειας πρέπει να τύχει μεγαλύτερης αναγνώρισης όσον αφορά την αξία του και τα κεφάλαια που ταπανώνται. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν ενέκρινε ένα ανακοινωθέν σχετικά με το αηφόρο, την αηφόρο ανάπτυξη και την υδατοκαλλιέργεια στόχος είναι πρώτον να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα υδατοκαλλιέργεια. δεύτερον να διατηρηθεί η βιώσιμη, ο βιώσιμο χαρακτήρα του και τρίτον να ε, βελτιωθεί η διακυβέρνηση του τομέα εισαγωγικά, η διαχείρισή του ίσω. Εδώ ε, πρέπει να ληφθούν μέτρα ε, σε όλα τα επίπεδα, από τι δημόσιες αρχέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που πλήττουν τον τομέα, για να στηρίξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια καλλιέργειας συμπεριλαμβανομένης και της ε, παραγωγής οστρακόδερμων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ε, την σχετική νομοθεσία σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι για να ορίσουμε προδιαγραφές για προϊόντα ε, και για οστρακόδερμα ε, τα οποία είναι αντικείμενο διεθνού εμπορίου. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει ένα εργαστήριο για ασθένειες ε, των μαλάκιων υπάρξει συντονισμών ε, των εθνικών εργαστηρίων και να υπάρχει επίσης και υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να ελέγχει την αφύσικη θνησιμότητα την στα οστρακοειδή τα στρίδια, με συγχωρείτε, τα τελευταία χρόνια, κάτι ε, το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει να ερευνήσουμε. Όσον αφορά την ευρύτερη στρατηγική για τις υδατοκαλλιέργειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επενθυμίσει τη συζήτηση που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2010 με βάση την έκθεση που προετοίμασε ο κ. Γκουίντο Μιλάνα. Η Επιτροπή ε, εκτιμά ε, την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει την υδατοκαλλιέργεια και να την προβάλλει περισσότερο. Εξάλλου θεωρούμε ότι οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει πρέπει να στηρίζονται μέσα από την κοινή ελευτική πολιτική και το στοιχείο αυτό πρέπει να ε, καλύπτεται κάτω από τη μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο τη μεταρρύθμισης τη κοινή ελευτικής πολιτική. Η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι πρέπει να βοηθήσει τον τομέα να οργανωθεί αποτελεσματικότερα. Ε, πιο συγκεκριμένα επιθυμούμε να ενισχύσουμε ε, τους παραγωγούς και τι διακλαδικές οργανώσει, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλότερη αξία των προϊόντων τους από το σωστό μάρκετινγκ και την σωστή επισήμανση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την πολύ περιεκτική απάντησή σας ε, και θα ήθελα να πω ότι σε μία πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία τα ψάρια ε, πολλές φορές είχαν λάθος ετικετοθυσία. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι έτρωγαν λάθος ψάρι και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Το γνωρίζει αυτό και πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι βραχυπρόθεσμα. Εκτός βέβαια από το να στηρίξουμε την ε, ε, υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ σημαντική και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε. Και μία ερώτηση από τον κύριο Γκάλαχερ. Πρόεδρε, χαίρομαι που άκουσα από αυτά που μας είπε η κυρία Δαμανάκη ότι η υδατοκαλλιέργεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η κοινή αληφτική πολιτική. Επίσης, θα ήθελα να πω στην κυρία Επίτροπο ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στην υδατοκαλλιέργεια κυρίως στις περιοχές όπου παρατηρείται υψηλός ρυθμός ανεργίας. Η Κομισιόν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία, να ανακοινώσει τις απόψεις επιτροπής στα κράτη-μέλη και να πει το εξής στα κράτη-μέλη. Βεβαίως και μπορούμε να συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ποιότητα όσον αφορά τα προϊόντα μας, αλλά καλύτερα να υπάρχει ένας φορέας που να ασχολείται με την υδατοκαλλιέργεια και να μην είναι κατατμημένη ε, η υδατοκαλλιέργεια σε αρμοδιότητες διαφόρων θεσμών. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Κάλαχερ ότι έχουμε πραγματικά τεράστιες ευκαιρίες ε, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό και σκοπεύουμε στην πρόταση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ να συντάξουμε ειδικό κεφάλαιο για την υδατοκαλλιέργεια. Και φυσικά θέλουμε να εξασφαλίσουμε και εξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή χρηματοδότησης για την υδατοκαλλιέργεια. Θα ήθελα να ενημερώσω και τον κύριο Κέλλη ότι φυσικά γνωρίζουμε το πρόβλημα και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας για την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων μας. Γι' αυτό και έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο για την σήμανση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει συνθήκες θεμητού και ισότιμου ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο μεταξύ των δικών μας αλλιέων και των αλλιέων που παράγουν προϊόντα τα οποία κατόπιν εισάγουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Παίρνουμε στην ερώτηση 41 του κυρίου Τσουκαλά. Την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσουκαλά για την ερώτησή του, γιατί πραγματικά το θέμα αυτό είναι μείζονο σημασίας. Θα ήθελα να πω ρητά και κατηγορηματικά ότι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας δυστυχώς δεν έχει φτάσει ακόμη σε, σε απρόσκοπτη λειτουργία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. 35 διάμεσες πληρωμές ε, ε, που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν μόνο το 70%. 70%. Ε, το το 5% της συνολικής ε, καταχώρησης κονδυλίων. Και μάλιστα η ετήσια έκθεση δείχνει ότι μέχρι το τέλη του, μέχρι το τέλη του 2009 18,2% του συνολικού κονδυλίου του Ταμείου Αλίας ε, είχε αφιερωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ θεαρητικό. Βέβαια τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο ε, προγράμματα τα, της, του πρώτου άξονα αλλά και άλλους άξονες. Μόνο άξονας 4 για την αηφόρα ανάπτυξη σε, σε περιοχές που στηρίζονται στην Ελία υστερεί επειδή απαιτείται πολύ χρονοβόλα διαδικασία για την θέσπιση εταιρικών σχέσεων. Και ο λόγος για την κατάσταση αυτή περιλαμβάνει καταρχήν την καθυστερημένη υιοθέτηση του κανονισμού για το Ταμείο Αλίας, την καθυστερημένη επίσης υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, γιατί μερικές φορές τα επιχειρησιακά προγράμματα υιοθετήθηκαν μόνο στο δεύτερο εξάμεινο του 2008. Το τρίτο πρόβλημα στην, αφορά τη σύσταση των, ελέγχων, των προγραμμάτων διαχείρισης και ελέγχου, γιατί η έγκρισή τους είναι η προϋπόθεση για την αποστολή πληρωμών. Και τέλος, τα, οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης που χτύπησε και τον αλληλευτικό τομέα. Σε αυτή, σε αυτή τη φάση της εφαρμογής είναι να πούμε το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχει υλοποιήσει τους στόχους του. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες που θα τις λάβουμε στα τέλη του 2011 στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Είναι δύσκολο να επισημάνουμε τις βέλτιστες πρακτικές, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικά κονδύλια στη διάθεσή τους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Και μάλιστα τα κονδύλια αυτά αφορούν διαφορετικούς άξονες και δεν μπορούμε να ε, αξιοποιήσουμε τον τρόπο, να αξιολογήσουμε τον τρόπο απορρόφησης. Γιατί για τον άξονα 1 ε, που αφορά τον ε, αλευτικό στόλο είναι πολύ πιο εύκολο να απορροφηθούν τα κονδύλια. Και μάλιστα στην συζήτηση που οργανώθηκε από την Βελική Προεδρία για να διορθωθούν τα προβλήματα απορρόφησης και ιδιαίτερα το πρόβλημα της πρόσβασης στο κεφάλαιο, η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποιες ε, ε, μεθόδους όπως τη χρήση, την απλούστευση κάποιων διαδικασιών και την απλούστευση των διατυπώσεων. Στην επόμενη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου θα, εξεταστεί η δυνατότητα διευκόλυνσης ε, αυτών των μέτρων. Και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 δυστυχώς έχει καθυστερήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2010 οι πραγματικές πληρωμές ε, ανέρχονταν μόνο στα 5.600.000 ε, ευρώ, δηλαδή μόλις 2% των συνολικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ελίας. 2% είναι ελάχιστο ποσοστό. Και αυτή η δυσάριστη κατάσταση οφείλεται κυρίως σε προγράμματα που αφορούν την διαχείριση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και κάποιες καθυστερήσεις ε, των μέτρων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Φυσικά, ορισμένες καθυστερήσεις οφείλονται και στην χρηματοπιστωτική κρίση, ιδιαίτερα τα μέτρα του δεύτερου άξονα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας για το 2009 και η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες ε, που θα ικανοποιήσουν την περιέργεια και τα διάφορα σκέλη τη ερώτηση του κυρίου Τσουκαλά. Δύο συμπληρωματικές, από τον κύριο Τσουκαλά η πρώτη και από τον κύριο Κέλλη η δεύτερη. Επιτροπώ για την πλήρη απάντησή της. Δράτω με την της μια που αναφέρθηκε στη δεινή οικονομική κατάσταση και στην μάλλον μη πλήρη εφαρμογή των σχετιζομένων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίες να ε, επισημάνω ότι θα ήθελα να ξέρω αν για την πλήρη απαγόρευση αλλιευτικών εργαλείων όπως για παράδειγμα της βιτζότρατας αυτό θα ενέπιπτε στην παροχή αποζημίωσης για τους αλληλείς που θα χάσουν τη δουλειά τους ή εάν ε, σύμφωνα με τον κανονισμό θα μπορούσε να γίνει επέκταση της διετούς διάρκειας παρεκκλήσεως από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμων κοινωνικών συνθήκων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κέλλη, ευχαριστώ ξανά κύριε Επίτροπε. Ποια κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα για τις βέλτιστες πρακτικές ήταν μια ερώτηση. Εγώ διρωτώ με και ποια ε, κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα για τις χείριστες πρακτικές. Μπορείτε να πείτε και να μας δώσετε κάποια, κάποιους λόγους για θέσεις διαφορές ανάμεσα στους καλύτερους και τους χειρότερους. Πριν σηκωθείτε κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας πω συνάδελφοι ότι είναι η τελευταία απάντηση αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω στον κύριο Κέλλη καταρχήν. Οι χώρες που έχουν καλύτερα συστήματα για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση και έχουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους, μπορούν με πιο εύκολο τρόπο να απορροφήσουν τα κονδύλια. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Πρέπει να ομολογήσω ότι οι μεσογειακές χώρες, οι νότιες χώρες, έχουν μεγαλύτερα προβλήματα απορρόφησης. Επίσης, πολύ συγκεκριμένα, κύριε Τσουκαλά, να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ακόμα πιο ειδικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους πάντες, ούτω ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο απορρόφησης. Γι' αυτό σκοπεύουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να απλουστεύσουμε τους κανόνες σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων και γι' αυτό έχουμε και μια γραμμή χρηματοδότησης στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του αλληλευτικού ταμείου, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να διευκολύνονται στην απορρόφηση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα σας κύριε Τσουκαλά για τον καονισμό για τη Μεσόγειο, αποφασίσαμε ότι αυτός ο κανονισμός για τη Μεσόγειο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Από την 1η Ιουνίου πρέπει να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό. Δεν μπορούμε να πιστοχωρήσουμε. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε αυτόν τον κανονισμό, θα χρειαστούμε δύο ή τρία χρόνια χωρίς συστήματα, να τα περάσουμε χωρίς συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης. Θα τον εφαρμόσουμε λοιπόν τον κανονισμό. Έχω ήδη συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ε, και έχω εξηγήσει στις αρχές αυτές ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός αμελητή. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις για τα ειδικά εργαλεία που είναι πολύ βαριά για το περιβάλλον, πολύ δυσάρεστα, όλες αυτές οι διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν. Επίσης, από πλευράς μας θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, ε, όλα τα περιθώρια που δίνει ο κανονισμός ε, για το Ταμείο, για να τους δώσουμε κονδύλια για την αποζημίωση. Αυτό αφορά και τις βιτζότρατες και τις στράτες και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, αλληλευτικό εργαλείο. Θα πρέπει να μας δώσουν παραδείγματα συμμόρφωσης και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ούτως ώστε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια χρηματοδότησης για να τους δώσουμε την ευκαιρία να βελτιώσουν τα εργαλεία τους και να βελτιώσουν την επιλεξιμότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώνουμε την ώρα των ερωτήσεων με αυτή την απάντηση. Τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα τις απαντήσουμε γραπτώς πέρα της συνεδρίασης. Σταματάμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 9 η ώρα.